Καλημέρα σε όλους, καλημέρα συνάδελφοι. Καλώς και πάλι στην ε, επιτροπή μας. Περιμέναμε κάποια λεπτά πριν να αρχίσουμε, αλλά νομίζω ότι τώρα έφτασε η στιγμή. Πρώτα απ' όλα, να εγκρίνουμε τη μερίσια διάταξη, το σημείο 1. Υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές, τις οποίες θα σας ανακοινώσω το σημείο 3, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης, 20-21 Φεβρουαρίου, ανα, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Το σημείο 9 είναι ένα σημείο το οποίο αναβάλλεται, δέσμευση σχεδίμηση των προϊόντων κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση. Τα σημεία 12 και 13 αιτήσει των εισογητών επίσης αναβάλλονται. Θα ήθελα να σας αναγγείλω ότι θα κάνουμε σε δύο μέρη σήμερα συνεδρίες των συντονιστών. Μία στις 11 παρατέταρτο, το πρώτο μέρος δηλαδή, και κλεισμένα των θυρών. Μετά, αφού διακόψουμε σε 11 παρατέταρτο λοιπόν, θα κάνουμε στο 10.30 συνεδρίες συντονιστών και το απόγευμα το δεύτερο μέρος στις 3.30. Μετά το με σημεριανό γεύμα. Το σημείο 20, αντιπροσωπεία στην ε, Κύπρο, 6 και 4, 4 ε, και 4. Και ένα νέο σημείο προσθέθηκε στη Μυρίσια Διάτοξη αύριο το πρωί στις 9, στις 9 ακριβώς. Δηλαδή η ανακοίνωση και η έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Τώρα, το σημείο 23 επίσης προσχώρησε προξένη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προσία των Δικαιωμάτων. επίσης, αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση 7 Μαου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορώ να θεωρήσω ότι έχει εγκριθεί η μερίσια δεξιά. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα, ορισμό εισηγητών. Η κυρία Βίξτρομ από την ε, Άλντε είναι η συγγήτρια για την διατύπωση της οδηγίας για τις ε, συνθήκες εισόδου και διαμονής ε, από τρίτες χώρες. Ο κύριος Ένσιου, συνεισηγητής και η κυρία Σόμερ για τον ε, κώδικα που αφορά τα, το πακέτο που αφορά τα σύνορα στα πλαίσια της συνθήκης Σέγγεν. Έχει καλός. Περνούμε λοιπόν στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι το σημείο 4, η τρέχουσα κατάσταση των ενεξελίξη διοργανικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των νομοθετικών διαδικασιών. Το δικαίωμα πρόσβαση δικηγόρο κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά την σύλληψη. Έχουν γίνει και συνεχίζονται δια, διαπραγματεύσεις για την προτινόμενη οδηγία για το δικαίωμα πρόσβαση σε δίκαιο. Θα ακούσουμε την ε, δική μας εισηγήτρια, την κυρία Άννα Ελένα Αντωνέσκιου, που θα μας πει σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και θα μας πει και κάποια πράγματα για τον τριμερή διάλογο. Έχετε το λόγο κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο έλαβε χώρα ο 7 κατά σειρά τριμερής διάλογος στα πλαίσια της οδηγίας που έχει να κάνει με το δικαίωμα των ανθρώπων που συμμετέχουν σε ποινική διαδικασία, το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, καθώ επίση και το δικαίωμα επικοινωνία μετά τη σύλληψη. Γίνανε έντονε συζητήσει, αλλά καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι προσπάθειε που κατέβαλαν προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές λύσεις όσον αφορά πολλές πτυχές της πρότασης. Συζητήσαμε για διάφορα άρθρα τα οποία πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν. Ορισμένες πτυχές είναι κυρίως τεχνικής φύσης. Και σε τεχνικό επίπεδο θα πρέπει να εξετάσουμε τις πτυχές αυτές. Ωστόσο, υφίστανται κάποια άλλα σημεία για τα οποία θα πρέπει να γίνουν και περαιτέρω συζητήσεις. Θα ήθελα γενικά να αφαιρθώ στα σημεία εκείνα για τα οποία χρειαζόμαστε περαιτέρω διευκρινήσεις. Όσον αφορά τους μάρτυρες, τον ενεργό ρόλο του δικηγόρου. Ως προς αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εξασφαλίσει ότι ε, θα προβλέπονται συγκεκριμένες διατάξεις για τη συμμετοχή του δικηγόρου κατά τη διάρκεια της ποινική διαδικασίας και της ανακριτικής διαδικασίας και ότι θα γίνεται σεβαστό το δικαίωμα αυτό. Όσον αφορά τώρα τη στάση των κρατών μελών στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου, υπόθηκε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να έχουν οι συμμετέχοντες σε μια ποινική διαδικασία πρόσβαση σε μια ενημέρωση όσον αφορά το δικαίωμά τους να έχουν δικηγόρο. Επίσης γίνονται κάποιες συζητήσεις όσον αφορά τα άρθρα που έχουν να κάνουν με την ε, ενημέρωση τρίτων ατόμων μετά τη σύλληψη και την, ε, το δικαίωμα του κατηγορουμένου του υπόπτου να έχει επαφή με τα άτομα αυτά. Επίσης συζητάμε τα άρθρα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με την ε, άρνηση χρησιμοποίησης δικηγόρου, την παρέτηση δηλαδή από το δικαίωμα αυτό και συζητάμε επίσης τα άρθρα αυτά που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Περαιτέρω άρθρα επίση συζητούνται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και του εισηγητή. Σημεία τα οποία θα συζητηθούν και στο, στην επόμενη ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Ανάμεσα στα σημεία που θα συζητηθούν είναι η παρέτηση από το δικαίωμα χρησιμοποίησης δικηγόρου, καθώς επίσης και κάποιες ε, παρεκκλήσεις όσον αφορά το δικαίωμα αυτό για γεωγραφικούς λόγους και επίσης θα συζητήσουμε και το ζήτημα της εμπιστευτικότητας των επικοινωνιών των συνομιλιών μεταξύ του υπόπτου, κατηγορουμένου και δικηγόρου. Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες αυτή τη στιγμή προκειμένου να ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Εκτιμώ ιδιαίτερα τις προσπάθειες της Ιρλανδικής Προεδρίας και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό για μας είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων αυτών. Να καταλήξουμε δηλαδή σε ένα κείμενο το οποίο θα εγγυάται προς τους ε, κατηγορουμένους ή στους υπόπτους ένα σαφές δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο και δικαίωμα επικοινωνία μετά τη σύλληψη, σύμφωνα με αυτά τα οποία ισχύουν σε διεθνέ επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου και με στη διάθεσή του για περαιτέρω ερωτήσει ή παρατηρήσει. Εδώ είμαστε σε, μια, σε ένα στάδιο που εξετάζουμε. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις καθώς και τα δικαιώματα. Έψαξα να σας βρω, κυρία Γκάντς. που έχετε και εσείς ε, συμμετάσχει πραγματεύσεις. Κάντε μας λοιπόν μια ενημέρωση παρακαλώ. Είχαμε έναν ε, πολύ επικοδομητικό διάλογο όλα τα μέρη. Το τελευταίος γύρος έγινε την ε, Δευτέρα. Κάποια ζητήματα εκρεμούν. Το πιο δύσκολο είναι η πράξη ε, κατά εξουσιοδότηση. Τα αναβάλαμε και ελπίζουμε να βρούμε μία λύση την επόμενη φορά στις 13 Μαΐου Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που εκκρεμούν. Πώς θα ενταχθεί η χάρτα στους συγκεκριμένους στόχους. Μιλάμε επίσης ε, για το μίσος και τις μειονοτικές ομάδες ή άτομα. Ε, επίσης τη διακριτική μεταχείριση και το πρόγραμμα ΕΠΣΚΙ και το πρόγραμμα καταναλωτών και κάποια εκτιμώντας το καλύπτουν. Ελπίζω λοιπόν να τελειώσουμε στις 13 Μαΐου. Να έχουμε μια έτοιμη πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκόντς για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Περνάμε στο τρίτο σημείο που αφορά τον κύριο Μέλο, εισηγητή για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας. Πείτε μας. Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να πω ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο θέμα, οι εργασίες εξελίσσονται ικανοποιητικά. Ήδη έχει υπάρξει συμφωνία κατά τη διάρκεια των τριμερών ε, διαλόγων σε σχέση με τα άρθρα 4, 1, 4 και 5. Στις 16 Απριλίου έλαβε χώρα η τελευταία συνάντηση και επιτεύθηκαν οι συμφωνίες που αφορούν ε, το ένταλμα έρευνες καθώς και όλα τα σχετικά θέματα. Υπάρχουν ακόμη άλλα άρθρα επίσης τα οποία ε, συζητήθηκαν και θα τύχουν συμφωνίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, συνεργασία του όλους τους σκιώδους εισηγητές, σκιώδεις με συγχωρείτε εισηγητές, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχαμε, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν οι σωστές αξιολογήσεις και να ληφθούν αποφάσεις. Διότι από τη μια έχουμε την διασφάλιση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και από την άλλη θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ε, διεξαγωγής αυτών των ερευνών με τρόπο σωστό και αποδοτικό. Ευχαριστώ λοιπόν και ελπίζω ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε αίσιο τέλος σε σχέση με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι τρεις εισηγητές λοιπόν μας έκαναν αυτή την ενημέρωση. Θα συνεχίσουμε αργότερα και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια η κυρία Ναταλή Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίδετε το λόγο. Με ευχαρίστηση σήμερα σας παρουσιάζω την έκθεση που αφορά την κατάσταση των ε, ανηλίκων και την πρόταση η οποία κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό εξάλλου αποφασίσαμε να συντάξουμε και γνωμοδότηση δεδομένου ότι κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά από τρίτες χώρες ή απάτριδες εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω δε ότι δεν ξέρουμε καν πόσος είναι ο ακριβής τους αριθμός. Έρχονται λοιπόν ασυνόδευτοι αυτοί οι ανήλικοι στην Ευρώπη και πριν να συναντήσουμε φορείς, εκπροσώπους, δημοσίου, αφού συνάντησα πάρα πολλούς ε, φορείς και εκπροσώπους ε, δημοσίων αρχών επιτόπου, να σας πω περιληπτικά ποιο είναι το περιεχόμενο της έκθεσης την οποία φαντάζομαι ότι όλοι έχετε λάβει στη μετρική σας γλώσσα και στρέφεται γύρω από δύο βασικές αρχές που θα χρησιμοποιήσω και ως μέθοδο για να σας αναλύσω το πρόβλημα. Πρώτη αρχή, η προστασία των παιδιών και όχι ο έλεγχος της μετανάστευσης, προστασία των παιδιών πρέπει να είναι εδώ η κινητήρια δύναμη. Το, η πρώτη αυτή αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ανήλικος είναι ένα ευάλωτο άτομο, ένα παιδί, το οποίο εισέρχεται στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ακόμη μια πιο λεπτή αρχή όσον αφορά την ε, εφαρμογή της σε νομικό επίπεδο. Θα πρέπει να υπερισχύσει το δικαίωμα, το θεμελιώδες του παιδιού. Είναι πιο λεπτή αυτή η έννοια, δεδομένου ότι ο ορισμός της χρησιμοποιείται και από την ομολογία και θα ήθελα να συμφωνήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε εμείς αυτό το ανώτερο συμφέρον του παιδιού να το ορίσουμε. Πριν να περάσω στις επόμενες παρατηρήσεις μου θα πω το εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει όχι μόνο τις πολλαπλές καταστρατηγήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών που διαπιστώνουμε, αλλά κυρίως τα κενά τα οποία υπάρχουν σε θέματα προστασίας των ανηλίκων. Και αυτό είναι ο στόχος της έκθεσής μου. Αυτό αιτιολογεί την δράση μας και τις απαιτήσει μας. Δεδομένου ότι όλοι συμφωνούμε, και αυτό είναι κάτι το είδαμε πάρα πολλές φορές και κυρίως στην Επιτροπή μας, ότι θα πρέπει σε θέματα προστασίας και συνθήκων υποδοχής η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ακόμη περισσότερο, να εξασφαλίσει τα ελάχιστα εχέγγυα ώστε να γίνονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών. Ποια είναι η πρώτη διαπίστωση στην οποία καταλήξαμε και πρέπει να ενεργήσουμε, έχουμε να κάνουμε με διάφορες διατάξεις κατακαιρματισμένες και διαφορετικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν ε, τα ανήλικα παιδιά. Σε κείμενα πρόσφατα, σε πιο παλιά, στο πακέτο για το άσυλο, στην ε, οδηγία. E Θα πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να φτιάξουμε εμείς ένα ε, μικρό οδηγό στον οποίο με απόλυτη ευκρίνεια και ευανάγνωστα να υπάρχουν όλες αυτές οι βασικές αρχές. Δεύτερη διαπίστωση, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. μια ιδεατή κατάσταση, ένα ειδικό ε, υποχρεωτικό εφαρμογής μέτρο για όλους θα ήταν πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι έχοντας εργαστεί για αυτό το θέμα του συναδέλφους, να ζητήσουμε ακόμη μία οδηγία, η οποία θα είναι δεσμευτική. Δεν είναι ίσως η κατάλληλη κατάσταση, διότι θα συνοδεύεται από ένα σύνολο μέτρων τα οποία ήδη υπάρχουν σε άλλα κείμενα. Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε στρατηγική σημασία κατευθυντήριε γραμμέ ώστε να έχουμε ένα ευέλικτο και εύκολα χρησιμοποιήσιμο μέσο από τις αρχές των κρατών μελών, τις αρμόδιες, που θα μπορέσουμε να φτιάξουμε αρκετά γρήγορα, σύντομο και τι προτείνω. Τις στρατηγικές γραμμές αυτές να τις παρουσιάσουμε ως ένα οδηγό κινούμενοι από τις βέλτιστες πρακτικές, από προδιαγραφές, από ελάχιστους κανόνες εφαρμογής για διάφορα σημεία κλειδιά. Κατά την άποψή μου αυτό το μέσον θα είναι πιο ρεαλιστικό, πιο συγκεκριμένο, πιο πραγματιστικό από μία κάποια στρατηγική, δεδομένου ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αποτελεί αυτή ήδη μια καποια στρατηγικη δεδομενου οτι το σχεδιο δρασης της επιτροπης αποτελει αυτής ηδη μια στρατηγικη γι' αυτό θα ήθελα να εγώ έχω ένα συγκεκριμένο μέσο, εύκολο, πρακτικό και χρησιμοποιήσιμο, πιο απλά. Για να μην μακρηγορήσω, έχετε αυτές τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές στην έκθεσή μου, Ποια είναι τα σημεία προτεραιότητας. Πρώτα απ' όλα το διεθνέ δίκαιο, καθώ και το ευρωπαϊκό, οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στο υπέρθετο συμφέρον των παιδιών. Αυτό όμως, αυτός ο ορισμός δεν έχει οριστεί και προτείνω βάσει κάποιων δικτών εμείς να μπορέσουμε να το ε, κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Βάση κάποιων αρχών που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο έχει κάνει η ΕΕ είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ώστε να αποτελέσει τη βάση για να φτιάξουμε αυτό το σύνολο δικτών. Δεύτερον, το περίπλοκο και ακαθόδες θέμα του καθορισμού της ηλικίας. Έχουμε μία σειρά παραδειγμάτων την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησης διάφορων στοιχείων ε, κάπως διεισδυτικών ιατρικών εξετάσεων που χρησιμοποιούν κάποιες χώρες για να καθορίσουν την ηλικία των νέων. Κατά την άποψή μου όμως, θα πρέπει να θεσπίσουμε μία κοινή ουμανιστική μέθοδο καθορισμού της ηλικίας. δηλαδή κριτήρια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και να σεβαστούν τα κρατη για να κάνουν τον καθορισμό της ηλικία. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να είναι μία ε, σειρά κριτηρίων πολλαπλών που να καθορίζονται από έναν εξάρτητο φορέα για να καθοριστεί η ηλικία των νέων. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αξιολόγηση αυτή. Κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ, την επίλυση αυτού καθόλου θέματος, είναι αυτό της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Υποστήριξης για το άσυλο, που έχει κάνει εργασίες πάρα πολύ στοχευμένες και θα μπορούσε να μας συνδράμει στο έργο αυτό και όχι μόνο σε αυτούς που ζητούν άσυλο. Επίσης, το θέμα των guardians, των κηδεμόνων. Κάθε χώρα θα πρέπει να θεσπίσει έναν υπεύθυνο ενήλικα από τη στιγμή που ο ανήλικας φτάνει στην επικράτειά του και ζητώ εδώ στην Επιτροπή να θεσπίσει κοινά πρότυπο όσον αφορά την εντολή, αρμοδιότητες και προσόντα του εν λόγω ατόμου αυτού του κηδεμόνου. Είδαμε ε, στο βελγικό παράδειγμα ότι υπάρχει ένας εξαιρετικός τρόπος που ακολουθείται και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πρότυπο. το σημείο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σέβονται και να εγγυώνται τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα των ανηλίκων. Όποια και αν είναι αυτά τα παιδιά και να αυτοί οι ανήλικοι να χαίρουν των ιδίων δικαιωμάτων που χαίρουν και οι ανήλικοι ε, υπήκοοι της χώρας στην οποία φτάνουν. Να έχουν ε, το κατάλληλο κατάλημα, την κατάλληλη ε, πρόσβαση σε θέματα παιδείας, υγείας. Πριν να επαναπροωθηθούν ή να ενταχθούν. Επίσης, το θέμα της ενηλικίωσης. Τα 18. Είναι ορόσημο για τα παιδιά. Και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει ένα ελάχιστο κατόφλι εναρμόνισης όσον αφορά τα εξατομικευμένα σχέδια περαιτέρω ζωής για τους ανήλικους. Ανάλογα με την κατάσταση του καθενός. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω, Πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο θέλω να κάνω αυτή την έκθεση γνωμοδότησης που πρέπει να είναι σύντομος παρά το γεγονός ότι στην αρχή διαφώνησα, τελικά συμφώνησε. Διότι πρέπει κανείς επιγραμματικά να πει. Και θέλω να πω τα κύρια σημεία και να τα εκφράσω με συγκεκριμένο τρόπο. Στις τελευταίες ανταλλαγές απόψεων, πολλές φορές είπα ότι η ισχύ αυτής της έκθεσης είναι ότι θέλουμε να καταλήξει σε ένα σύντομο κείμενο και όπως λένε και οι Γερμανοί, ούκαν το πολλό το F περίπου. Πρέπει κανείς να είναι σύντομος αλλά περιεκτικός. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει ε, υποχρεωτικά να κάνω θα μας οδηγήσει στο να έχουμε ένα σύντομο κείμενο ε, πρακτικού περιεχομένου, χωρίς πολλά μπλα μπλα, για να του προσδώσουμε την ισχύ που θέλουμε. Και βεβαίως είμαι σίγουρη ότι με την συνεργασία σας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μια τέλεια εκθέση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους βοηθούς, καθώς και τη γραμματεία που πραγματικά εργάστηκαν ε, με πάρα πολύ ε, σωστό τρόπο και ενεργητικά ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την έκθεση που θα είναι τιμή για όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκίσμπεκ. Αρχίζουμε με τις συνεισηγητές Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, Νάταλη. Είναι χαρά η συνεργασία μαζί της. Συμφωνώ με τις γενικές αρχές. Δηλαδή το παιδί είναι πρώτα απ' όλα παιδί και μετά μετανάστης. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα καλύτερα, τα συμφέροντα του παιδιού πρώτα απ' όλα. Και μετά να γίνει η ατομική αξιολόγηση. Τώρα για να γίνουν συγκεκριμένοι και να περάσουμε στα πρακτικά, γιατί όλα τα άλλα έχουν υποθεί. Θεωρώ πως πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στα κράτη-μέλη παρά στην ε, Κομισιόν, υπό την έννοια πως ε, όταν βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη, συχνά υπάρχει ε, η νομοθεσία, αλλά η εφαρμογή είναι διαφορετική μεταξύ των κρατών μελών. Τον τελευταίο μήνα συνάντησα όχι μόνο αρχές, ε, οργανώσεις, ε, συμβούλια μετανάστευσης, δήμους κτλ. αλλά και ασυνόδευτούς ανηλίκους που ε, ήρθαν στη Σουηδία. Η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι η χώρα στην Ευρώπη που καλωσορίζει τους περισσότερους, υποδέχεται τους περισσότερους ασυνόδευτους ανηλίκους. Και αναμένουμε το 2013 γύρω στους 4.000. Το 2012 ήταν 1.500. Ε, είναι λοιπόν μεγάλη πρόκληση. Όταν ε, μίλησα λοιπόν... Ναι, κάποια παιδιά τα οποία είναι στην Σουηδία εδώ και λίγα χρόνια από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Σομαλία οι ιστορίες τους ήταν συγκινητικές και θα σας πω το βασικό πρόβλημα. Ταξιδεύουν 6-7 μήνες, πέρασαν από το Ιράν, από την Τουρκία, από διάφορες χώρες και δεν ήξεραν πού είναι. Έφτασαν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, σε άλλες χώρες και όταν έφτασαν στη Σουηδία βεβαίως επικρατούσε το καθεστώς του Δουβλίνου για το οποίο ε, δεν είχαν καμία ιδέα και ήταν ένας εφιάλτης. Ε, κρατώντας ε, κάποια κράτη-μέλη που δεν πίστευε κανείς πως θα ε, είχαν παιδιά υποκράτηση, αλλά είχαν κρατηθεί. Οπότε η αβεβαιότητα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η έλλειψη πληροφοριών, το γεγονό πως τους έστελναν μπρος πίσω, μπρος πίσω και τελικά έπαιρναν άσυλο ή άδεια παραμονής στην Σουηδία και το καλό σου ήταν πως ε, έμπαιναν στο σχολειο αμεσω αμέσως μετά από τρει-τέσσερι μέρες ε, γράφουν στο σχολείο. Και αυτό στα μάτια τους ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνονται δηλαδή πως ε, είχαν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν. Οπότε τι λέω Ναταλή. Είναι η διαφορά που υπάρχει στην εφαρμογή μεταξύ των κρατών μελών. Όχι για λόγους κακής πίστης, επειδή δεν υπάρχουν πόροι, δομές, εκπαίδευση. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές, γιατί πολλά συμβαίνουν, ε, πολλά πράγματα έχουμε ψάξει, να δούμε τι γίνεται. Οπότε αναρωτιέμαι μήπως ε, μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για αυτόν τον κατακαιρματισμό που αναφέρετε για να βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Και μετά επίσης θα πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε, που είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης Ασύλου και τη Frontex. Γιατί το λέτε κι εσείς ε, στην έκθεσή σας για τη συλλογή των δεδομένων που είναι μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο για άσυλο, γιατί δεν ξέρει κανείς αν θα ζητήσουν άσυλο ή όχι. Ε, τα παιδιά που έρχονται στις χώρες μας. Ε, η Frontex ήδη συλλέγει δεδομένα, της χάρη. Θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε κάποια δεδομένα. Η πατιαρμοστία του ΟΗΕ έχει μια καλή βάση. Μετά, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να αφαιρθώ σε κάποια σημεία του κειμένου. Ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που βασίζεται σε κάποιους δείκτες νομίζω είναι πάρα πολύ καλή πρόταση. το θέμα της αύξησης του συντονισμού με τρίτες χώρες πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποια πιλωτικά έργα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Το ζήτημα των συγκεκριμένων τίτλων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Μετανάστευσης, ειδικά για τους ανηλικούς, γιατί πρέπει να διατεθούν τα λεφτά. Επίσης, η Κομισιόν να υιοθετήσει δεσμευτικές ε, κατευθυντήριες γραμμές. Τι εννοείς εδώ πέρα δεσμευτικές. Επίσης το να μην κρατείται ποτέ ο ανήλικος. Ε, εδώ πέρα νομίζω αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή. Το ζήτημα των περισσότερων πληροφοριών σε μια γλώσσα και μορφή που μπορούν να καταλαβαίνουν. Χαίρομαι που μπορώ να πω πως στο πακέτο του ασύλου που πέρασε έχουμε βάλει μια τέτοια τροπολογία και αξίζει να τη στηρίξουμε. Το θέμα του Κίδεμόνα δεν ξέρω αν η Κομισιόν πρέπει να ορίσει κοινέ προδιαγραφέ. Μπορούμε να δούμε τι υφιστάμενε βέλτιστες πρακτικές. Επίσης το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην υγεία, πολύ επίμαχο θέμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τελειώσουμε κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το πακέτο του ασύλου. Όταν προτείνουμε να εξαιρούνται πάντα από την επιταχυμένη διαδικασία, κάτι το οποίο είναι ένα θέμα εξαιρετικά επίμαχο. Και τελικά το απέρριψε το Συμβούλιο και μετά προτείνουμε το αρμόδιο κράτος θα πρέπει πάντα να είναι αυτό το οποίο, ε, στο οποίο έγινε η πιο πρόσφατη αίτηση ασύλου. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Οπότε, εκτός αν ξανανοίξει όλη η συζήτηση για το άσυλο, γιατί θα ψηφιστεί το πακέτο του ασύλου τον Ιούνιο και ξέρετε πως ήταν πολύ σοβαρή διαπραγματευσία. Αν τα ανοίξουμε λοιπόν αυτά τα δύο θέματα, ε, πρέπει να ξανανοίξουν όλες τις διαπραγματεύσεις του ασύλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ Νόταλη. Κύριε Κοράτσα, δεν ήθελα να σας διακόψω, αλλά πρέπει να σας υπενθυμίσω πως έχουμε αρκετούς σκιώδες συζητητές και έχουμε 10 παρατέταρτο ψηφοφορία, οπότε τα ίδια θα γίνουν. Δηλαδή, ανυπόμονοι βουλευτές ε, έρχονται στις 9.45 για την ψηφοφορία και έχουμε δύσκολη ψηφοφορία για τα στοιχεία αεροπορικών επιβατών. Οπότε μην ξεχνάτε πως 10 παρατέταρτο πρέπει να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Κύριε Τζίπελ. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οι δύο συνάδελφοι ανέφεραν αρκετά σημεία, οπότε μπορώ να είμαι σύντομη. Να ευχαριστήσω την Νάταλη Γκρίσμπεκ γιατί ε, το θέμα είναι σημαντικό αλλά και πολύ πολύπλοκο, αυτό αναφέρθηκε ήδη, γιατί ήδη για το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων υπάρχουν υπάρχει κάποια συζήτηση και για τα ιδιαίτερα δικαιώματα του παιδιού. Και εδώ πέρα υπάρχουν κάποια έγγραφα, οπότε η πρόκληση πραγματικά είναι να δούμε τις διαφορετικές διατάξεις που υπάρχουν και το... εάν έχουμε και διαφορετικές διά... μεγάλες διαφορές πραγματικά εντός των οδηγιών και βεβαίως το ζήτημα της ιδιαίτερης προστασίας του παιδιού και το πώς αξιολογείται κάθε φορά. Αλλά νομίζω πως η συγγήτριά μας εδώ πέρα βρήκε μια πάρα πολύ καλό τρόπο να κάνει προτάσεις, να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές, πώς έχει εφαρμογή στα κράτη-μέλη, τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Και να δούμε πού πρέπει να δράσουμε, είτε πρόκειται για νέες οδηγίες, είτε για περισσότερα ερεθίσματα. Απλά να σας υπενθυμίσω πως ανεξαρτήτως του γιατί κατέληξε ένα ασυνόδευτος ανήλικο σε κάποιο κράτο μέλο και ανεξαρτήτω του στάτου που έχει το ζήτημα τη πρόσβασης ε, στην εκπαίδευση νομίζω θα μπορούσε να είναι ε, κεντρικό και νομίζω πως ε, μπορούμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό ιδιαίτερος και νομίζω πως έχουμε εδώ πέρα μια καλή βάση για την περαιτέρω εργασία. Λοιπόν, η κυρία Φλότρ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω και εγώ κάποια λόγια για την έκθεση αυτή, γιατί θεωρώ ότι η πρόταση που γίνεται από την εισηγήτριά μας πραγματικά συνάδει με τις βασικές μας ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων αυτών ατόμων, δηλαδή των παιδιών, των ασνόδευτων ανηλίκων και ότι λαμβάνονται υπόψη το υπέρτατο συμφέρον τους σε κάθε απόφαση η οποία θα λαμβάνεται. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια επιμέρους σημεία της έκθεσης που πιστεύω ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμα και σε κατάθεση τροπολογιών. Πολλά πράγματα είπαμε και έχουμε δίκιο κάθε φορά που μιλάμε για όλες αυτές τις διαφορετικές υποχρεώσεις και τις διατάξεις που υφίστανται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, δικαίου αλλά ξέρετε ότι υπάρχει έπειτα και η νομολογία όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους και ιδίως όσον αφορά την εξέταση του υπέρτατου συμφέροντών τους. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια τελογική σκέψη σχετική, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όντως θα λαμβάνεται υπόψη η βασική αυτή αρχή, όπως άλλωστε το εξήγησε και η συγγήτρια. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τι ακριβώ θα ζητήσουμε με την έκθεση αυτή. Έχει δίκιο και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ όταν λέει ότι ε, πρέπει να δούμε πόσο δεσμευτικέ μπορεί να είναι αυτέ οι στρατηγικέ κατευθυντήριε γραμμέ. Σίγουρα λέμε ότι ε, μολονότι θέλαμε μια οδηγία, η οδηγία δεν ήταν ρεαλιστική και ούτε μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Επομένω βρισκόμαστε μεταξύ οδηγία και κατευθυντήριων γραμμών. Το σημαντικό είναι η ε, νομική μας βάση να μπορεί να ισχύσει στα κράτη-μέλη, αν μπορούμε να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές με σημεία επαφή εθνικά, με εθνικά σχέδια δράσης, με συγκεκριμένες τακτικές ημερομηνίες αξιολόγησης αυτών των ε, σχεδίων, των εθνικών σχεδίων δράσης, μήπως τελικά η εναλλακτική αυτή είναι η καλύτερη δυνατή μέθοδος εργασίας και συντονισμού Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως αυτή θα ήταν η κατάλληλη λύση για να εξυπηρετήσουμε τους στόχους μας. Και να πούμε επίσης ότι θέλουμε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων να μετασχηματιστεί σε task force, γιατί όπως είπαμε το δικαίωμα των παιδιών εμφανίζεται σε πάρα πολλούς τομείς της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε τη δημιουργία, τη θέσπιση μιας task force, η οποία να ασχολείται ακριβώς με το ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε ήδη βασιζόμενοι στην Επιτροπή των Επιρογνωμών να δημιουργήσουμε μια task force. Όσον αφορά τώρα την επιστροφή, όσον αφορά τους ανήλικους οι οποίοι ετούνται άσυλο, διακόπτει ο Πρόεδρος. Κυρία Φλότρα, σας παρακαλώ πολύ. αναφέρομαι σε όλου αυτού που μπαίνουν τώρα στην αίθουσα. Υπάρχει ένα συνάδελφό ο οποίο ομιλεί αυτή τη στιγμή. Καθίστε, αλλά μην κάνετε θόρυβο, παρακαλώ πολύ. Ετοιμαστείτε για την ψηφοφορία. Σεβαστείτε όμω τον συνάδελφό ο οποίο μιλάει αυτή τη στιγμή. Κύριε Φλότρα, σα δίνω το λόγο. Ναι, σα έλεγα λοιπόν ότι όσον αφορά του ανήλικου ετούντε άσυλο, όλα αυτά διευθετούνται στο πακέτο ασύλου μέσω των διαφόρων μεσών που έχουμε εκεί. Θα πρέπει ε, λοιπόν να συμφωνήσουμε με την εισηγήτρια ότι θα πρέπει σε μια κοινή δέσμη μέτρων να καλύψουμε όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τους ασνόδευτους ανηλίκους που ετούνται άσυλο. Τώρα όσον αφορά την επιστροφή υπάρχουν πολλές παράγραφοι στην έκθεση. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των παραγράφων αυτών. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε ότι η αξιολόγηση της οδηγίας για την επιστροφή που θα γίνει φέτος θα μπορούσε να ασχοληθεί συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει δηλαδή αυτό, με το ζήτημα της επιστροφής των ασυνόδευτων ανηλίκων. Δηλαδή μέσω της αναθεώρησης και της εξαιολόγησης ενδιάμεσης οδηγίας για την επιστροφή να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Και βέβαια ένα άλλο σημείο για το οποίο η νομολογία είναι πάρα πολύ σημαντική είναι πάρα πολύ σημαντικό η επιστροφή να λαμβάνει και αυτή η χώρα στα πλαίσια του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού και θα πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ρήτρε διασφάλισης, τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση και ενδεχομένω θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ακόμα και στην επαγγελματική εμπειρία, την επαγγελματική άσκηση, ακόμα και πριν την ηλικία των 18 ετών, είναι πιθανό για πάρα πολλού ανηλίκου να καταφέρουν να έχουν πρόσβαση σε μια κάποια επαγγελματική πείρα που θα καταφέρει κατά αυτόν τον τρόπο να εμπλουτίσει τη μετέπειτα ζωή του. Αυτά είναι τα βασικά μου σημεία, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο τροπολογιών. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή με τόσο θόρυβο στην αίθουσα. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν δείξτε ένα κάποιο σεβασμό μη τι άλλο προς, τον, προς συναδέλφους οι οποίοι παίρνουν το λόγο. Σας ευχαριστούμε κυρία Φλότρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μπρόγκς, θα σας ακούσουμε και εσάς, αλλά στη συνέχεια ας ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή από ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πολλά ζητήματα να ψηφοφορήσουμε, αρκετά πολύπλοκες ψηφοφορίες αυτή τη στιγμή. Επομένω, ας ολοκληρώσουμε γρήγορα, σας παρακαλώ πολύ. όσα μέλη βρίσκονται στην αίθουσα, σας κάνουν ησυχία και το ίδιο, το ίδιο αίτημα απευθύνω και προς βοηθού οι οποίοι δίνουν αυτή τη στιγμή στου βουλευτέ του, του κατάλογους ψηφοφορία. Κύριε Μπρόγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο, ε, όσο και η προλαλή σα. Μα λέτε πω πρέπει να προηγούνται τα δικαιώματα του παιδιού. Να προηγούνται από, του, από, ε, από τι. Αλλά βεβαίως δεν ε, είναι σωστές και δεν συνηθίζονται οι ολόκληρες προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω ε, αυτό το εννοούμε με υλικού όρου. Δηλαδή το παιδί θα τραφεί καλύτερα και θα είναι πλουσιότερο από ότι αν ήταν στον τρίτο κόσμο. Όμω πρόκειται για μια εθνοκεντρική υπόθεση εδώ πέρα. Δηλαδή το παιδί στην Ευρώπη χωρίς ρίζες και χωρίς ε, πολιτισμική υποστήριξη είναι προτιμητέο από το να ζει στη χώρα του. Βεβαίω, εάν είναι προτιμητέο, πρέπει λογικά να θεωρηθεί πως κανένα παιδί δεν μπορεί να ζει στον τρίτο κόσμο. Εμείς σήμερα στην Λίμπε πρέπει να πάμε στην Αφρική και όπως η Μαντόνα, η τραγουδίστρια ας πούμε, να απάγουμε και να φέρουμε στην Ευρώπη όποιο παιδί δούμε. Βεβαίως η ιδέα πως τα παιδιά θα έχουν τους πόρους, τη γνώση και ε, τα μέσα να έρθουν μόνα τους ε, στην Ευρώπη είναι κάτι το φανταστικό. Αν έρθουν ασυνόδευτα σημαίνει πως έχουν πέσει θύμα τράφικινγκ είτε από εγκληματίες είτε από τις οικογένειες και τους γονείς τους ή Ε, βεβαίως από αυτούς που εφευρίσκουν τις φοβερές αρχές ε, που ακούσαμε εδώ πέρα που θα προσελκύσουν ως μαγνήτης ολόκληρο τον πληθυσμό του τρίτου κόσμου. Αυτοί οι λαθρέμποροι ανθρώπων δεν ανησυχούν πραγματικά για τα δικαιώματα των παιδιών, είναι πιόνια στο παιχνίδι και το παιχνίδι βεβαίως είναι να αλλάξει δημογραφικά ο πληθυσμός της Ευρώπης και να υπάρξει εθνική εκαθάριση των αυτοχθόνων πληθυσμών. Ευχαριστώ και ελπίζω να ήμουν σύντομος. Μάλιστα. Η Κομισιόν. Ε, παρακαλώ να είστε σύντομος. Ναι, θα είμαι. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκρίσμπεκ για την έκθεση που συμφωνεί και με δικές μας ανησυχίες που είναι στο μεσοπρόθεσμο μεσοπρόθεσμη έκθεση και στο πρόγραμμα δράσης. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις συστάσεις. Απλά φάνηκε νομίζω συζήτηση πως έχει μεγάλη σημασία να συνδεθούν όλοι οι φορείς που ασχολούνται με τους ασυνόδευτους ανηλίκους π.χ. το θέμα του Κιδεμόνα στην Ολλανδία και αυτοί θέλουν να έρθουν σε επαφή με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες ακριβώς για να μην υπάρχουν προβλήματα και κενά στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αλλιώς, γενικώ θα ήθελα να πω πως θα είμαστε σε επαφή με το γραφείο της κυρίας Γκρίσμπεκ. Επίσης ε, έχουμε και εμείς κάποιες ερωτήσεις για το τι εννοούμε με τις δεσμευτικές ε, στρατηγικές κατευθυντήρες γραμμές και θα θέλαμε να μάθουμε πώς κατέληξε σε αυτή τη διατύπωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Κομισιόν, τους βουλευτές, τους σκιώδης Δεν έχουμε πολύ χρόνο για περαιτέρω συζητήσει, αλλά βεβαίω η κυρία Γκρίσμπεκ, η συγγήτρια, ε, μπορεί να ολοκληρώσει. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, κάπως ηλεκτρισμένο κλίμα, για να μην πω σε αταξία τελειώνει η συζήτηση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και την Κομισιό που με βοήθησαν και για την σύνταξη της έκθεσής μου. Όντως θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την συνεργασία. Θα ήθελα... Πω, πω, πω. Δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν ε, θα επαναλάβω όλες τις υποδείξεις, παρατηρήσεις και σχόλια των συναδέλφων. Τους ευχαριστώ, τις σημείωσα. Υπάρχουν πολλά σημαντικά στοιχεία, όντως κυρίως το θέμα της ε, αξιολόγησης, από την ε, οδηγίας επιστροφής η βοήθειά σας όσον αφορά τους τρόπους τους οποίους θα γίνει η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι παρατηρήσεις της Αναμαρία που ξεκινάει από το πρώτο που γνωρίζει καλύτερα και την κατάσταση που γνωρίζει καλύτερα, την κατάσταση στη χώρα της, αλλά δεν είναι η συνήθις κατάσταση στην Ευρώπη. Και στην έκθεσή μου Είπα ότι ίσως στον ευρωπαϊκό χώρο έγκυται να ανεβάσει τον πύχη για να έχουμε μια σφαιρική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι πάρα πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομη, σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις συνεργασίες μας και όταν κατατεθούν οι τροπολογίες, τύπης και ουσία, θα προσπαθήσω να κάνω την τελική μου έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ κυρία Γκρίσμπερ. για, τις, ε, για τα αποτελεσματά σας. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 6 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τα μέλη και πάλι. Παρακαλώ. Προσοχή. Για την ψηφοφορία έχουμε πολύπλοκα θέματα. Σας υπενθυμίζω πόσο σημαντικό είναι να βρείτε την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας και να τη χρησιμοποιήσετε σωστά. Να τις έχετε έτοιμες τις κάρτες. Και αρχίζουμε με την πρώτη έκθεση. Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες των ναρκωτικών. Αρχίζουμε. Ησυχία παρακαλώ στην αίθουσα. People in the room who are not voting, at least remain in silence. Παρακαλώ, όσοι δεν θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, σιωπήσουν τουλάχιστον. Λοιπόν. Getting started. Αρχίζουμε. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογίες που θα ψηφιστούν on block. Πρόκειται για την 22, 25, 26, 28, 31, 36, 42, 44. On block λοιπόν, τις ψηφίζουμε on block. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 6 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 30 χωρίζεται σε δύο μέρη. Ψηφίζουν το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση του δευτέρου μέρους τροπολογίας 30 παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. «28 προς 26 εγκρίνεται». «29 υπέρ». «Κατά». «Αποχές εγκρίνεται». «7». «Καταπίπτει». «Όχι». Την ψηφίζουμε. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 7 ζητείτε. Κυρία Ματίας, τι θέλετε. Επαλήθευση της 7. Εντάξει λοιπόν. Θα ψηκα... ηλεκτρονική ψηφοφορία της 7. Ε, 7. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ήρεμα, δεν θέλω πανικό, λέει ο πρόεδρο. Αρχίζει ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. 22 υπέρ 33 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 ηλεκτρονική επαλήθευση της 34 αρχίζει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία 29 προς 26 εγκρίνεται 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10 καταπίπτει. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Καταπίπτει. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται CA1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 μία, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε τώρα το κείμενο έτσι όπως το τροποποίησαμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 46 προς 3 και 5 αποχές. Ευχαριστούμε κυρία Χέντ. Τώρα θα περάσουμε το επόμενο θέμα το οποίο αφορά την ε, διαπραγματευτική ομάδα και την ε, συμφωνία τους. Ευχαριστούμε κυρία Χέγκ. Περνούμε τώρα στην ε, πολιτική έγκριση της συμφωνίας τη οποία επέτυχε ο εισηγητής και οι συνεισηγητές ε, η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του τριμελούς διαλόγου της 21ης ε, Μαρτίου η συγγήτρια η κυρία Σιλβί Γκυλιόμ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη η ψηφοφορία. 44 υπέρ, 3 κατά. 8 εποχέ. Προχωρούμε. Ευχαριστούμε κυρία Γκυγιόμ. Στο Eurodac τώρα. Δημιουργία του συστήματος Eurodac. Η κυρία Μακοβέη, η συγγετρία. Τελική ψηφοφορία για το τελικό κείμενο. Αρχίζει η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. 42 προς 8 και 5 αποχές. Ευχαριστούμε κυρία Μακοβέη. Περνούμε τώρα. Τελευταία ψηφοφορία που είναι και η πιο εκτεταμένη και η πιο πολύπλοκη ας πούμε. Συγκεντρωθείτε λοιπόν παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Χρήστε δεμέ περίπτωση επιβατών αφορούν το περίφημο PNR. Ο εισηγητή είναι ο κύριος Τίμωθη Κίρκοπ. Θέλετε να κάνετε δήλωση πριν από την ψηφοφορία. Ε, πρόεδρε, όχι τόσο δήλωση. Δράτω με τις ευκαιρίες που έχει ο εισηγητής ε, να κάνει μερικά σχόλια πριν την ψηφοφορία κυρίως επί της διαδικασίας. Με ακούτε? Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως δεν χρειάζεται νομίζω να υπογραμμίσω στην Επιτροπή τη σημασία της συγκεκριμένη οδηγίας. Την ε, διαδικασία που έχουμε περάσει της συζήτησης, τον ανοιχτό και διαφανή τρόπο με τον οποίο ελπίζω ότι λειτουργήσα για όλες τις ομάδες και τις ε, γνωμοδοτήσει και μάλλον δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω πως το βλέπω εγώ, δηλαδή ως κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. 16 κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή έχουν ή σχεδιάζουν ένα δικό του σύστημα πληροφοριών αεροπορικών επιβατών. Οπότε είναι σημαντική αυτή η οδηγία για να έχουμε ένα συνεπές ε, σύστημα στην Ευρώπη συνολικά και Επίσης, δεν νομίζω πως χρειάζεται να υπενθυμίσω σε κανέναν το τι ακούσαμε από τους ειδικού για τις επιτυχίες που είχε το σύστημα αυτό στην καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας ε, και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό το ζήτημα. Θα ήθελα εδώ πέρα να ευχαριστήσω το προσωπικό μου, το προσωπικό όλων των μονίμων αντιπροσωπιών στις Βρυξέλλες που με βοήθησαν πάρα πολύ στη διαδικασία αυτή τους ε, εμπειρογνώμονες που μίλησαν και κατέθεσαν τις διαφορές υπηρεσίες που ήρθαν εδώ και σε όλα τα μέλη των ενδιαφερομένων ομάδων ε, τους και οδησίγητες και όλους τους υπολείπους και του ε, επί της διαδικασίας της σημερινής ψηφοφορίας. Πρώτα απ' όλα θα ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα που έχει υποβληθεί για να απορριφθεί αυτή η πρόταση. Οπότε θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καταψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα και μετά θα περάσουμε στην ε, κύρια ψηφοφορία και βεβαίως για λόγους ε, συνεκτικότητας ε, έχουμε χωρίσει την ψηφοφορία σε μπλοκ. Έχουμε το μπλοκ από 1 έως 7 που αφορά τρομοκρατικές ενέργειες, το δεύτερο αφορά τρομοκρατικές ενέργειες και διασυνοριακά εγκλήματα, το άλλο αφορά τις πτήσεις, το τέταρτο αφορά τις διεθνείς πτήσεις, ε, το πέμπτο ενδοευρωπαϊκές, ε, το έκτο αφορά ένα ε, σύστημα ε, επέκτασης, ε, ένα κεντρικό σύστημα PNR και ένα σύστημα προαιρετικό. Οπότε, οι 4 και οι 5, εάν υιοθετηθεί η 5 ε, κατά τη 5 και 6 και 7 πάνε μαζί επίσης ε, και θα έχουμε δύο τελικές ψηφοφορίες ε, πρώτα απ' όλα στο τροποποιημένο κείμενο και μετά για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων και θα ήθελα να ζητήσω κύριε Πρόεδρε να ψήσουμε με ηλεκτρονική κάρτα ειδικά την πρώτη ψηφοφορία για το ψήφισμα που στόχο έχει την απόρριψη της πρότασης. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την συνεισφορά σας. Thank you, thank you, Mr. for your, for your... Ευχαριστούμε κύριε Κυρκόπ για τις διευκρινήσεις αυτές όσον αφορά την πολυπλοκότητα, την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα της ψηφοφορίας που μόλις τώρα θα κάνουμε. Ξέρετε ότι δεν είναι μόνο σημαντικό το ζήτημα ως προς την ουσία του, αλλά υπάρχει και αυτή η πολυπλοκότητα προς τον τρόπο ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες και το τροποποιημένο κείμενο και ψηφίζουμε και για την έναρξη διαπραγματεύσεων. Καθώς επίσης και για τη διαπραγματευτική ομάδα. Δεν υπάρχουν συμβαστικές τροπολογίες αυτή τη φορά. Επομένως, θα ψηφίσουμε, όπως είπε ο εισηγητής on block, ομαδικά. Θα έχουμε μια πρώτη ψηφοφορία ως προς την απόρριψη της πρότασης και στη συνέχεια θα έχουμε κάποιες ψηφοφορίες όσον αφορά τα διαφορετικά μπλοκ, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, συγκεκριμένες πτήσεις, είδος πτήσεις, είδος συστήματος. Και το καθένα ανταποκρίνεται στη διαφορετικό μπλοκ τροπολογιών. Μπλοκ 1, μπλοκ 2, μπλοκ 3, μπλοκ 4, 5 και στη συνέχεια έχουμε την έκτη και την έβδομη ομάδα τροπολογιών, μπλοκ 6 και μπλοκ 7. Ας συγκεντρωθούμε λοιπόν προτάθηκε από τον εισηγητή μας τον κύριο Κίρκχοπ να ψηφίσουμε χρησιμοποιώντας την ε, κάρτα μας, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά δηλαδή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι με την αρχική ψηφοφορία, ουσιαστικά δηλαδή με την τροπολογία 36, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Δύο μέλη του ΕΛΚ επιπλέον υπάρχουν. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Κοιτάξτε λίγο, συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δύο επιπρόσθετες ψήφοι. Μπορείτε να κάνετε κάτι. Μία ψήφος επιπλέον αυτή τη στιγμή ακόμα. Εντάξει, το λύσαμε το πρόβλημα. Για να δοκιμάσουμε πάλι. Τι έχουμε, για να δούμε. 30 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Εντάξει, τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε. Δεν ήταν τελικά τόσο πολύπλοκο. Κυρία Ματιέ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ πολύ συνάδελφοι. Ναι, να πούμε ότι μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τη ψηφοφορία αυτή δεσμεύεται για την καταπολέμηση τρομοκρατίας. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για πολύ σημαντική ψηφοφορία. Δεν ψηφίζουμε τίποτα το σοβαρό και νομίζω ότι θα πρέπει να αποτίσουμε φορό τιμή στα άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους στην Βοστόνη. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι θύματα της τρομοκρατίας και δεν είμαστε σοβαροί. Μετά από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι το λόγο. Κύριος Βέμπερ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Το αποτέλεσμα δεν πήγε όπως θα ήθελε το ΕΛΚ. Θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία του θέματος. Όλοι ξέρουμε πως είναι σημαντικό το θέμα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο, τους ε, συντονιστές ε, και τους υπόλοιπους να σκεφτούν αν υπάρχει κάποια δυνατότητα να γίνει αυτή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Πρέπει να δούμε αν γίνεται να μην συζητηθεί μόνο εδώ πέρα, αλλά να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, να μπορέσουν να αποφασίσουν όλοι οι βουλευτές και να αντιμετωπίσουν τις ερωτήσεις στις χώρες τους. Και ζητάω τι τις υπηρεσίες ε, να μου απαντήσουν στο ερώτημα αυτό, γιατί νομίζω πως ε, είναι πραγματικά απαραίτητο να διεξαχθεί αυτή η ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το δείτε. Second. Mrs. Interveld. Η κυρία Νιτφέλτ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρώτα απ' όλα δε, θα ήθελα να διαβεβαιώσω το ΑΕΛΚ πως όλοι και αυτοί που υπερψήφισαν αυτές τις τροπολογίες ε, είναι υπέρ της καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας και της ασφάλειας όλων των πολιτών μας. Αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να πει κανείς πως απορρίπτοντας αυτή την πρόταση δεν θέλουμε την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως η πρόταση αυτή έχει υποβληθεί με διάφορες μορφές ε, ε, εδώ και 7 χρόνια είναι ένα επίμαχο ζήτημα. Εγώ προσωπικά ως κοιόδη συγγήτρια έχω προσπαθήσει να πείσω τον εισηγητή να περιμένει μετά την ε, έγκριση τη οδηγία προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων γιατί νομίζω πως συνδέονται τα δύο ζητήματα και ελπίζω γρήγορα να εγκρίνουμε αυτή την οδηγία και μετά να συζητήσουμε αυτή την πρόταση. Εγώ δεν ήθελα να τεθεί σε ψηφοφορία αλλά ε, αυτή τη στιγμή σε τέθη και επέμεναν οι άλλες ομάδες αυτό ήταν το μόνο δυνατό αποτέλεσμα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρη πως θα επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με νέα πρόταση. Ελπίζω να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί εδώ και πολλά χρόνια στο Κοινοβούλιο και μετά να μπορέσουμε επιτέλους να συμφωνήσουμε σε ένα σύστημα που θα μας ικανοποιεί όλους. Κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω την ευαισθησία της κυρίας Μπεσερίλ σε σχέση με το θέμα αυτό της τρομοκρατίας, αλλά εκπλήσωμαι που δεν ήταν η σχέση της που μίλησε εξ ονόματος του ΕΛ και ότι πρόκειται για πολιτική θέση. Εγώ θα αιτιολογούσα το σύστημα αυτό του PNR για την τρομοκρατία και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ εκθέσει εκ μέρους της Επιτροπής που λέγει ότι δεν μας χρησιμεύει το θέμα του PNR για την καταπολέμηση τρομοκρατία. Άρα δεν είναι επίγον να το εγκρίνουμε τώρα. Εάν πρόκειτο ε, για κάτι το επίγον και το χρήσιμο, θα το κάναμε, θα το εγκρίναμε. Αυτό αφορά άλλου είδους ε, εγκλήματα ή παραπτώματα τα οποία αφορούν φερρυπίν, την κράτηση, άλλου τέτοιου θέματα ποινικού περιεχομένου. Θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό υπέψη. Και έτσι το συζητήσαμε. Με αυτή την πολιτική δεν έχει κανένα, ε, καμία λογική τη στιγμή κατά την οποία ακόμη συζητούμε την οδηγία και τον κανονισμό να εγκρίνει μια τέτοια εξουσία με το PNR. Καταλαβαίνω τη δική σας ευαισθησία, συνάδελφε, αλλά σύμφωνα με την Επιτροπή αυτό το μέσο δεν είναι έγκαιρο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο θέμα του PNR. Ευχαριστώ. Κύριε Κίρκοπ, κύριε Πρόεδρε, η δική μου αντίδραση είναι η ακόλουθη, όχι απογοήτευση, όχι μόνο απογοήτευση, αλλά βλέπω ότι υπάρχει και υποκρισία, πολύ μεγάλη υποκρισία. Μου φαίνεται πραγματικά παράδεκτο να ακούω αυτές τις παρατηρήσεις από την κυρία Ινβέλτε, η οποία αυτή τη στιγμή χειρίζεται το φάκελο που έχει να κάνει με το καναδικό PNR, και ελπίζω ότι θα εγκαταλείψει τουλάχιστον την εργασία αυτή. Γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο μας λέει είναι ότι εμείς κάνουμε κάποιες συμφωνίες με το PNR, με τις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής, με τον Καναδά, με την Αυστραλία και ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε εμάς τους ίδιους, να έχουμε το δικό μας ευρωπαϊκό PNR στην Ευρώπη. Επομένως, τι είναι το τόσο θετικό με τις υπόλοιπε αυτές χώρες και για ποιο λόγο δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε και τα ίδια, να έχουμε τα ίδια πρότυπα εδώ στην Ευρώπη. Θέλουμε να έχουμε πραγματικό έλεγχο και πραγματική ασφάλεια για τους πολίτες μας στην Ευρώπη. Με την απόρριψη αυτή πηγαίνουμε πίσω χρόνια, οπισθοχωρούμε. Και όχι μόνο αυτή τη στιγμή θα έχουμε 16 απλώ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που θα κάνουν ό,τι θέλουν χωρί να υπάρχει κανένα έλεγχο, αλλά το ίδιο πράγμα θα μπορούσαν να κάνουν και οι υπόλοιπε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντα εντελώ διαφορετικέ μεθόδου πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν προστατεύει κανέναν στην Ευρώπη, ούτε αυτούς οι οποίοι επισκέπτονται τις χώρες μας. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη κατάσταση, απέσια πραγματικά. Και δεν θα με πείραζε αν πραγματικά οι συνάδελφοι είχαν κάποιε ανώτατε αρχέ, τι οποίε έπρεπε να σεβαστούν. Αλλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι χρησιμοποιούνται ψευδή επιχειρήματα προκειμένου να δικαιολογηθεί η δηλία πολλών συναδέλφων, η έλλειψη θάρρου για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Είμαι ιδιαίτερα αναστατωμένο και ενοχλημένο σήμερα και έχω κάθε λόγο να είμαι ενοχλημένο από τη στάση των συναδέλφων και από το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή μα αντιμετωπίζει με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο αυτή την έκθεση. Ούτε λέξη πλέον δεν θέλω να ακούσω για τις δίθεν αυτές αιτιολογήσεις ότι κάνουμε δίθεν το καλύτερο για τον Ευρωπαίο πολίτη και περιμένουμε πρώτα να εγκριθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι να περιμένουμε να εγκριθεί πρώτα το Ευρωπαϊκό Σύστημα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων δεν μας εξυπηρετεί καθόλου, γιατί ουσιαστικά δεν θα καταφέρναμε να εγκρίνουμε γρήγορα το σύστημα αυτό. Το θέμα είναι να μπορούσαμε εμείς στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι να εγκριθεί το σύστημα αυτό, να έχουμε τα απαραίτητα πρότυπα για το PNR. Ενδεχομένω να χρειαστεί να περιμένουμε 3, 4, 5 και 6 χρόνια μέχρι να έχουμε το σύστημα για τα προσωπικά δεδομένα. Σε όλο αυτό το διάστημα, πάρα πολλά ευάλωτα άτομα θα πλήττονται από εγκληματικέ ενέργειες, από τρομοκρατία και το καθεξής. Πραγματικά δεν μπορούμε να εργαζόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε χάσει ουσιαστικά την βασική ιδέα του καθήκοντος που εξυπηρετούμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι η κυρία Εντιβέλτ πρέπει να εγκαταλείψει την έκθεση την οποία επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή με τα PNR του Καναδά και να τη δώσει σε κάποιον άλλον. Η δήλωσή της είναι καθαρά υποκριτική για μένα. Σας παρακαλώ πολύ λίγη ησυχία, κύριε Όλμπρεχτε. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Έχει ζητήσει πρώτο το λόγο. Σας ζητώ συγγνώμη. Όλμπρεχτ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις για το σύστημα αυτό. Για πάνω από ένα χρόνο συζητάμε την πρόταση αυτή και όπως ξέρετε εμείς οι πράσινοι έχουμε απορρίψει τα συστήματα PNR και τις συμφωνίες PNR εξ ολοκλήρου γιατί θεωρούμε ότι η διατήρηση των δεδομένων αυτών, τα συστήματα profiling που χρησιμοποιούνται δεν συνάδουν με τα συνταγματικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συνάδουν με την ε, νομολογία πολλών εθνικών δικαστηρίων, αλλά και με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Η πρόταση για ένα ευρωπαϊκό PNR έχει πλέον απορριφθεί. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στην Ευρώπη δεν είναι σημαντική. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα, Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνα. Εργαζόμαστε για μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για το τι σημαίνει κίνδυνος το τι σημαίνει ύποπτο πραγματικά κριτήρια και όχι θεωρητικά κριτήρια για έναν θεωρητικό κίνδυνο ή συστήματα παρακολούθηση οποιοδήποτε πολίτη εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιοδήποτε κράτο. Αυτό ακριβώ θέλαμε να αποφύγουμε. Αυτό το γενικό κλίμα υποψία που θα βάρινε όλε τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλαμε να αποφύγουμε. Λάβαμε μια πολιτική απόφαση στην Επιτροπή μα και αυτή την πολιτική απόφαση πρέπει να τη σεβαστούμε τώρα. Εμεί πάντα λαμβάνουμε αποφάσεις εδώ χωρίς κανείς να αφισβητεί την ε, νομιμότητα των αποφάσεων αυτών. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση αυτή. Μην προσπαθήσετε τώρα να παρακάμψετε μια απόφαση η οποία είναι σαφής, είναι πολιτική, εκπροσωπεί την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής μας και την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων που κατέριψαν, απέρριψαν την πρόταση αυτή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες ευκαιρίες στο μέλλον για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, ακόμα και με τα δεδομένα των επιβατών αν δούμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της στο Βοστόνη ή άλλα συμβάντα, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες υπήρχαν διαθέσιμε πληροφορίε Οι άνθρωποι αυτοί που έκαναν στρομοκρατικές ενέργειε στη Βοστόνη ήταν ύποπτοι και στο παρελθόν υπήρχαν για αυτούς πληροφορίες. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή εμεί να συσσωρεύουμε όλο και περισσότερε πληροφορίε για του μη υπόπτου. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη διαστοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για του ήδη φυστάμενου υπόπτου. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να βελτιώσουμε. Και θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πρότυπά μα για να καταλήξουμε σε μια κοινή βάση και αυτό να αποτελεί προπόθεση για καλύτερη και πιο βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως και το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς επίσης και την αρχή του κράτους δικαίου κάθε φορά. Ας σεβαστούμε λοιπόν την απόφαση που μόλις τώρα πήραμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω εντελώς με τον Τίμωθη Κέρκοπ και είμαι απογοητευμένος για το ότι δεν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια ενιαία ρύθμιση για την Ευρώπη. Σήμερα υπερψηφίσαμε έναν κατακαιρματισμό στην Ευρώπη, το οποίο δεν είναι καλό για τους ε, πολίτες. Εγώ θα ήθελα η ε, απόφαση αυτή να μεταφερθεί στην Ολομέλεια και όσοι ε, λένε πως πρέπει να περιμένουμε οποιοδήποτε άλλο θέμα, δεν ε, ισχύει κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη αλλάζουν, τα συστήματα αλλάζουν συνεχώς. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε συνεχώς στην ε, επικαιρότητα. Νομίζω αυτό αποδείχτηκε σήμερα. Δεν έχει δηλαδή κανένα νόημα να περιμένουμε άλλα πράγματα. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο για να μην έχουν διαφορετική αντιμετώπιση οι πολίτες. Εδώ πέρα μπορούσαν πραγματικά να κάνουμε κάτι για να ξέρουν και οι πολίτες πού βρίσκονται και να μην χρειάζεται κάθε φορά να σκέφτονται ε, μήπως ε, στη χύψη χώρα αποθηκεύονται, ξέρω εγώ, στη Μεγάλη Βρετανία 10 χρόνια τα δεδομένα. Είχαμε μια ευκαιρία να τα περιορίσουμε στα 3 χρόνια, ε, την οποία τη χάσαμε. Ας ακούσουμε τώρα έναν δεύτερο γύρο. Ε, δύο βουλευτές θέλουν να δευτερολογήσουν να απαντήσουν σε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Και μετά και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να... Η κυρία Χιμένες Βεθερίλ. Θα ήθελα να απαντήσω στην ε, κυρία Κάρμεν Ρομέρο το εξής. Ίσως δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπα δεν ήθελα να πω ότι αυτοί που καταψήφισαν την έκθεση δεν είναι κατά, κατά πολέμης της τρομοκρατίας. Το ξέρω, ξέρω ότι όλοι επιθυμούμε να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό που είπα είναι ότι θεωρώ ότι είναι έλλειψη σεβασμού. Αρχίζοντας την ε, ψηφοφορία να κάνουμε κάτι αντίθετο με αυτό που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο είναι η προστασία των πολιτών. Ας κάνουμε τα πράγματα πιο με πιο σοβαρό τρόπο. Χάσαμε μια ευκαιρία. Και εγώ είπα ότι θα πρέπει τα πράγματα να τα κάνουμε σεβόμενοι τους ε, πολίτες. Δηλαδή, ψηφίζουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ενεργήσαμε είναι σωστός. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν δυσαρεστηθεί που δεν προχωρήσαμε στην έγκριση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Η κυρία Ινβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, στον κύριο Κίρχοπ, που θέλει να μου κλείσει το στόμα, δεν θέλει να με ξανακούσει, να πω ότι δυστυχώ είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω το δικαίωμα, όπω όλοι, να λαμβάνω το γράμμα. Με κατηγορείτε ότι είμαι υποκρίτρια βάσει λανθασμένων γεγονότων. Θα θυμάστε ω συγγήτρια για την, ε, ε, το θέμα του PNR, είπα Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπληκτική. και δεν θυμούμε όταν έχασα την ψηφοφορία αυτή να είμαι τόσο κακιά ως ιτημένη όσο τώρα. Δεν θέλω να υπερψηφιστεί το θέμα του PNR και η συμφωνία με την Αυστραλία, όχι γιατί με ενδιαφέρει και είμαι φαν του θέματος, αλλά αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι εδώ να αντικατοπτρίσουμε στις εκθέσεις αυτές την θέση του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω με τον Καναδά να παρετηθώ. Θα δω ποια είναι η τη της Επιτροπής μας. Θα δω ποιες συζητάσεις που θα κάνω. Δεν ξέρω αν θα υπέρ ή θα καταψηφίσω. Και όπως και εσείς και εγώ έχω το δικαίωμα να εκφράζω την απόψή μου. Γι' αυτό κύριε Βός επίσης δεν πιστεύω ότι πρόκειται για ατύχημα. Νομίζω ότι είμαστε συνεκτικοί ευθύ εξ αρχής. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πότε είχα πει ότι θα υπερψηφίσω το θέμα αυτό και μετά να με κατηγορήσετε ως υποκρίτρια. Πάντα εγώ ήμουν συνεκτική με αυτό που έκανα. Ήθελα να καταλήξω σε συμβιασμό, αλλά είπα ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υιοθετηθεί η οδηγία για την προστασία δεδομένων. Δεδομένου ότι αυτό είναι η βάση της συνεργασίας ε, αστυνομίας δικαστικών ερχών στα θέματα αυτά. Εάν λοιπόν θέλουμε να κατηγορήσουμε αυτούς οι οποίοι υπερψήφισαν την πρώτη ε, τροπολογία ότι δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, αυτοί είναι οι υποκριτές. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η κατηγορία. Now, Mrs. Κύριε Χολμάιερ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αντιλαμβάνομαι τον Τίμωθη Κέρκχοπ ε, και λόγω εμπειρίας ε, ως ε, Υπουργός Εσωτερικών τώρα. Για αυτό το οποίο λέει η κυρία Λόπες πως δεν προσθέτει τίποτα αυτό. Βλακίες. Όχι βεβαίως ότι το PNR λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά είναι ένα συστατικό κομμάτι στην όλη προσπάθεια καταπολέμησης τρομοκρατίας και των χειρότερων μορφών της. Άνθρωποι υφίστανται βλάβεση και πεθαίνουν γιατί δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για να δράσουμε προληπτικά. Και, κυρία Ινετφέλτ, εγώ νόμιζα πως ε, ο κύριος ε, Κέρκοπ ε, εννοεί πως είστε υποκρίτρια γιατί λέτε πως ε, είστε υπέρ του συστήματος PNR ενώ δεν ήσασταν ποτέ. Τώρα το να μας λέτε πως εξαρτάται από την προστασία των δεδομένων κτλ. Με συγχωρείτε, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Εξαρτάται απλά από το τι θα ορίσουμε εμείς από κοινού. Αυτό το οποίο ε, λέτε σημαίνει πως δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε επαρκώς την τρομοκρατία. Δεν θέλετε βεβαίως να αναλάβετε τέτοια ευθύνη, αλλά θα υπάρχει έλλειψη δεδομένων. Αν συμβεί κάτι λόγω πληροφοριών που δεν έχουμε, όμως θα πρέπει να υπομειστείτε αυτή την ευθύνη, είτε σας αρέσει είτε όχι. Αλλά αυτό το οποίο με ενοχλεί εμένα περισσότερο είναι πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμερίζει τον εαυτό του. Δηλαδή από μόνο του μπαίνει στο περιθώριο. Γιατί τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν μόνα τους διακυβερνητικά, χωρίς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υπογράψουν τις συμφωνίες τους. Οπότε, τι θα έχουμε. Σε, σε μια συμφωνία το 2020 τι δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί, γιατί δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε ε, με το Συμβούλιο, δεν θέλετε να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, ενώ κατέβαλε πραγματικά προσπάθειες ο κύριος Κέρκοπ. Εντάξει, σεβαστή η απόφαση, αλλά εδώ πέρα πρέπει μετά ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Αλλήμον, δεν λέω πως δεν θέλετε να καταπολεμήσουμε την ε, τρομοκρατία, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Αλλά το πώς θα γίνει αυτό και πόσο ε, αυστηροί θα είμαστε σε αυτό, δεν συμφωνούμε. Προφανώς το ΕΛΚ ε, θέλει μια πιο αυστηρή και στιβαρή πορεία στο θέμα αυτό. Και για αυτά τα οποία είπε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, Πράγματι είναι λογικό νομίζω να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, να ρωτήσουμε ολόκληρη την Ολομέλεια, να δούμε αν συμφωνεί ολόκληρο το Κοινοβούλιο με αυτήν εδώ πέρα την άποψη. Δηλαδή να κάνουμε συμφωνίες με Αυστραλία, με ΙΠΑ και να μην εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας. Κυρία Άνστ, επίσης ε, συγγήτρια. Ναι, ευχαριστώ. Μια αρχική παρατήρηση. Τώρα για τα χειροκροτήματα νομίζω ε, φτάνει για σήμερα, έτσι. Κοιτάξτε, ελήφθη μία απόφαση και ακριβώς για το σεβασμό της ασφάλειας των πολιτών και των θεμελιωδών τους ε, δικαιωμάτων, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, για τις διάφορες κατηγορίες που ακούγονται, δεν στέκουν. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω. Πρώτον, ελήφθη μία απόφαση, έτσι. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε εδώ πέρα. Πως τέσσερι ομάδες από την αρχή είχαν πει ξεκάθαρα πως το σύστημα όπως έχει καταρτιστεί ε, δεν θα μπορέσει να περάσει. Το είχαν πει σε όλες τις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Το λέγαμε συνεχώς. Δεν ήταν τυχαία αυτή η απόφαση. Δεν είναι όπως τα λέτε. Μήνες καθίσαν όλες οι ομάδες μαζί και πραγματικά ποτέ δεν υπήρξε μια πιστική απόδειξη για το ότι αυτό το σύστημα είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της θερμοκρατίας. Το πρώτο είναι αυτό και πρέπει να σας πω πως απορρίπτω και αυτό το οποίο ακούστηκε για την Σόφη Ινιτφελντ. Είναι άδικο να ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία και να, να μιλάτε έτσι για τη συνάδελφο. Να σας πενθυμίσω επίσης, είχαμε και πολλές συζητήσεις ε, ισχυώδης αλλά και εδώ πέρα, πώς χρειαζόμαστε πρώτα ένα κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων και να ρυθμίζει τα δικαιοσύνης και εσωτερικών και μετά μπορούμε να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Ξανά και ξανά επανήλθε η πρόταση Ε, να αποφασίσουμε πρώτα την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων και μετά να συζητήσουμε ε, ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών. Και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένας κανονισμός. Αλλά ένας κανονισμός. Όχι δύο και τρεις και να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Και είναι σαφής. Εάν απορριφθεί εδώ μέσα δεν μπορεί να πάει κάτι στην Ολομέλεια. Άμα δημιουργήσουμε τέτοιο προηγούμενο τότε θα λέμε ναι, έτσι θα το αποφασίσουμε εδώ και μετά αλλιώ ε, αλλού, ανάλογα τις πλειοψηφίες. Ελήφθη μία απόφαση, πρέπει να τη σεβαστούμε. Δεν έχουν πάντα δίκιο το ΕΛΚ και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί. Μάλιστα, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές ακόμα που θέλουν να τοποθετηθούν. Κυρία Σίπελ. Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την ε, Συμφωνία Πληροφοριών Αεροπορικών Επιβατών και την ε, καταπολέμηση τρομοκρατίας συχνά είναι μια έντονη συναισθηματική συζήτηση που απομακρύνεται από τα γεγονότα και φοβάμαι από το πώς εξελίσσεται η συζήτηση. Η κυρία Χολμάιερ στο τέλος της παρέμβασής της είπε πως δεν κατηγορεί κανέναν για το ότι δεν θέλει να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα είπε πως εμείς φέρουμε την ευθύνη, όσοι καταψηφίσαμε δηλαδή, εάν αύριο κάπου λάβει χώρα μια τρομοκρατική ενέργεια. Δηλαδή μια φοβερή δήλωση, ειδικά δεδομένων των ε, θυμάτων της ε, Βοστόνης, είναι πραγματικά θλιβερό να λέμε πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα δεδομένα, γιατί έχουν ένα τέτοιο σύστημα εδώ και καιρό οι Ηνωμένε Πολιτείε και παρόλα αυτά δεν εμπόδισαν αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Είμαι βαθύτατα πεπισμένη πως ε, η απόφαση αυτή δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα προστασίας δεδομένων, πράγματι, αλλά θεωρώ πως ήδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξετάσουμε το εάν είναι όντως πρόβλημα μίας ακόμα οδηγίας ή αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τι υφιστάμενε οδηγίες και να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των αρχών πριν ε, αποφασίσουμε περαιτέρω μέτρα. Η σημερινή απόφαση δεν είναι μία ε, ατομική απόφαση των βουλευτών. Υπήρξαν συστάσεις τεσσάρων κοινοβουλευτικών ομάδων να απορριφθεί αυτή η απόφαση. Και όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Βέμπερ, ενοχλούμε λίγο, έτσι για να το πω ήπια. Είτε υπάρχει ε, άρθρο στον κανονισμό που λέει πως όταν απορριφθεί μια οδηγία στην Επιτροπή πρέπει να πάει μετά στην Ολομέλεια ή δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο. Αν δεν υπάρχει τέτοιο άρθρο στον κανονισμό, είναι νομίζω αναξιοπρεπές να δημιουργήσουμε τέτοιο προηγούμενο και να λέμε μήπως με κάποιο κολπάκι μπορούμε να βρούμε κάτι για να το στείλουμε στην Ολομέλεια. Νομίζω ε, πρέπει να μην κάνουμε τέτοια πράγματα, να αποδεχτούμε την απόφαση που ελήφθη. Κύριε Βέμπερ, κύριε Πρόεδρε, επί της αλλά και πρώτα απ' όλα μια παρατήρηση επί της ουσίας γιατί η πλειοψηφία εδώ πέρα, η αριστερή πλευρά προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει. Γεγονός είναι πως η προστασία των δεδομένων των πολιτών μέσω της απόρριψης σημερινής θα επιδεινωθεί γιατί θα ισχύουν τα εθνικά συστήματα. Και σήμερα πραγματικά εξασθενήσατε την ευρωπαϊκή προστασία των δεδομένων. Τώρα, να έρθω στην διαδικασία. Σήμερα έχουμε, ε, είχαμε εδώ πέρα να ψηφίσουμε μία ε, έκθεση. Είχαμε μία νομοθετική πρόταση της ε, Κομισιόν. Και είχαμε μία έκθεση, αλλά ψηφίσαμε μόνο μία τροπολογία. Όχι ολόκληρη την έκθεση. Πρόκειται για μία μόνο τροπολογία. Θεωρώ λοιπόν πως πρέπει πρώτα απ' όλα να περάσουμε σε μια τελική ψηφοφορία επί της πρότασης Κομισιόν όπως αυτή τροποποιήθηκε, η οποία πρέπει να γίνει νομίζω στην Ολομέλεια. Και σας παραπέμπω στον κανονισμό, στο άρθρο 56, όπου λέει πως η απόρριψη νομοθετικών προτάσεων γίνεται στην ε, Ολομέλεια και στο άρθρο 196 επίσης λέει σαφώς πως οι επιτροπές δεν έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις της Κομισιόν. Εμείς λοιπόν ερμηνεύουμε τον κανονισμό ως εξής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε μια τελική ψηφοφορία επί της ε, προτάσεως Κομισιόν η οποία θα επιβεβαιωθεί στην Ολομέλεια. Και σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να ακολουθήσετε τον κανονισμό. Και την συζήτηση που κάνουμε εδώ πέρα να την κάνουμε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όλη η αριστερή πλευρά φοβάται ξαφνικά την Ολομέλεια. Εάν είναι ξεκάθαρες οι πλειοψηφίες όπως μας λέτε και αν όλοι οι συνάδελφοι των κοινοβουλευτικών ομάδων θα ψηφίσουν όπως ψηφίσατε εδώ πέρα σήμερα, δεν χρειάζεται να φοβάστε την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου εμείς είμαστε πεπισμένοι πως αυτά γράφει ο κανονισμός και παρακαλούμε να το ακολουθήσει αυτό και ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εξής κατάσταση. Θα ψηφίζαμε για μια μισή περίπου ώρα, ακριβώς επειδή προβλεπόταν ότι η ψηφοφορία θα ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη. Και είδαμε ότι ε, εγκρίθηκε ευθύς αμέσως η τροπολογία αυτή για την απόρριψη της πρότασης. Και στη συνέχεια ορισμένοι συνάδελφοι αποφάσισαν να κάνουν δηλώσεις, ο ένας μίλησε εναντίον του άλλου, κάποιοι έθιξαν κάποια ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία που ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι προτού απαντήσω στα σημεία αυτά θα πρέπει να ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Τώρα πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τη δυνατότητα να πάει η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια όπως ζητήθηκε. Ας ολοκληρώσουμε όμως πρώτα τον κατάλογο των ομιλητών, ας δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να πάρουν το λόγο και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα διαδικαστικά ζητήματα. Η κυρία Σαρτζεντίν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω καμία συζήτηση για την ψηφοφορία PNR, την οποία μόλις κάναμε, αλλά ως συντονίστρια για τους πρασίνους, άκουσα δηλώσεις από διάφορους συναδέλφους, οι οποίοι ουσιαστικά λένε ότι θα πρέπει να αγνοήσουμε εντελώ το ότι είχαμε μια δημοκρατική ψηφοφορία και άκουσα κάποιοι οι οποίοι αναφέρονται και σε διάφορα άρθρα του κανονισμού, σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να παρακάμψουμε το γεγονό ότι είχαμε μία ψηφοφορία εδώ που έχασε μία πολιτική ομάδα. Μπορεί να μην είμαι μέλο τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα εδώ, οπότε είμαι μαθημένη στο να χάνω που και που. Αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα σε μια δημοκρατία. Και πραγματικά με σοκάρει που μετά από μία ψηφοφορία διεξάγεται συζήτηση για το πώ θα παρακάμψουμε αυτή την ψηφοφορία διεξάγεται μια συζήτηση που ουσιαστικά εκβιάζει τους συναδέλφους οι οποίοι καταψήφισαν λέγοντάς τους ότι κάνανε, πήρανε μια πολύ λανθασμένη απόφαση. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι εξφεδονίζουν τέτοιες δηλώσεις δεν σέβονται το ίμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλους αυτούς οι οποίοι ψήφισαν για πολιτικές ομάδες όπως η δική μου πολιτική ομάδα, οι οποίοι πολύ προσεκτικά αποφάσισαν τι θα πρέπει να γίνει με τα δεδομένα PNR και το πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. θα ήθελα να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να συζητάμε σε ένα πνεύμα δημοκρατίας και φοβάμαι ότι αυτό το πνεύμα μας έχει εγκαταλείψει πια στην αίθουσα αυτή, σε αυτή την Επιτροπή. Πρόεδρος, ναι, κύριε Κύρκο, προφανώ εσεί έχετε το τελευταίο λόγο, αλλά σα ακούσουμε τον κύριο Πίκερ πρώτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παραβλέπουμε το εξή. Εδώ πέρα συνέβησαν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα νομίζουμε. Πρώτα απ' όλα, εδώ πέρα παριστάνετε πως θέλετε να έχουμε κοινέ προδιαγραφές, ενώ ε, τι θα γίνει, οδηγούμαστε στι εθνικές προδιαγραφές και δεν έχουμε τελικά ευρωπαϊκές. Και εμποδίσατε πολύ περισσότερα πράγματα από την χρήση των δεδομένων για την αποτελεσματική καταπολέμηση και πρόληψη της τρομοκρατίας. Εμποδίσατε και την χρήση των δεδομένων για την καταπολέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό ήταν το δεύτερο κομμάτι. Δεν εμποδίσατε μόνο την ε, επιτυχέστερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και τη χρήση αυτού του μέσου για την ε, οργανωμένη και βαριά εγκληματικότητα. Η Δανία ήδη έχει ένα καλό εθνικό παράδειγμα. 80% των εγκλημάτων ναρκωτικών ε, μπόρεσαν να εξηχνιαστούν χάρη σε αυτά τα δεδομένα. Υπάρχουν λοιπόν θετικά παραδείγματα από τα οποία φαίνεται πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δεδομένα. Έχετε λοιπόν διπλή ευθύνη και πραγματικά αμελήσατε το καθήκον σας για την εσωτερική ασφάλεια, για την ασφάλεια των πολιτών. Και πλέον φροντίσατε, όπως είπα, για την εσωτερική ανασφάλεια τελικά. Και αυτό είναι ευθύνη των αριστερών. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Θα είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε, να στηρίξω τον εισηγητή, τον κύριο Κέρκοπ και τους ε, συναδέλφους Μάνφρεντ Βέρμπερ και για το ζήτημα της ε, δυνατότητας ε, του να εκφραστούν όλοι οι συνάδελφοι στην Ολομελία. Αν το επιτρέπει ο κανονισμός, γιατί να μην το κάνουμε. Καθώς ε, δεν θέλουμε εμείς να παρακάμψουμε και να μην σεβαστούμε αυτά τα οποία λέει η Επιτροπή. Αν το συνδέσουμε, Σόφη, με την ε, προστασία των δεδομένων σημαίνει ότι νύπτουμε ως ε, πόντιος πιλάτος ασχήρας μας. Δεν θα κάνουμε τίποτα σε αυτή τη θητεία. Δεν προλαβαίνουμε. Ε, δηλαδή πατάτε και λίγο στο έδαφος, να είστε λίγο ρεαλιστές. Δεν θα το δούμε καθόλου το ζήτημα, θα περάσουν χρόνια. Στην επόμενη εντολή ξέρεις πως έχουν διαδικασίες. Στην επόμενη θητεία. Οπότε αν το συνδέσουμε με την προστασία των δεδομένων σημαίνει πως δεν θα κάνουμε τίποτα. Έτσι δίνουμε τις αρμοδιότητές μας μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνα, πίσω στα κράτη-μέλη. Οπότε θα πρέπει νομίζω να ε, ακούσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους στην Ολομέλεια. Ναι ή όχι. Όχι να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες. Μία ψηφοφορία ναι ή όχι στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα στον εισηγητή, στον κύριο Κύρκοπ. Πρόεδρε, Γίνονται διάφορα σχόλια ότι θέλουμε να παρακάμψουμε τους κανόνες. Αντιθέτως, εμείς τους ακολουθούμε. Θα ήθελα, παρακαλώ, εσείς με τον ε, υπάλληλο που ασχολείται με αυτό το θέμα, με που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, να δει ποιος είναι ο κανόνας διαδικασίας που ισχύει και τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δούμε... Ε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να το παραπέμψουμε το όλο θέμα στην Ολομέλεια, η οποία θα εγκρίνει ή θα απορρίψει το θέμα. Ας κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Πρώτα απ' όλα. Ακούσαμε κάποιες επεξηγήσεις ψήφου αυθόρμητα και έγιναν και κάποιες ε, δηλώσεις αλλά για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, νομίζω ότι είναι σωστό πούμε ότι συμφωνούμε εδώ όλοι ότι το θέμα που μας απασχολεί εδώ και το σημαντικό δεν είναι να πούμε αν είμαστε κάθετα αντίθετοι προς οποιοδήποτε μορφή τρομοκρατίας. Κανένας εδώ δεν μπορεί να θέσει ένα αμφιβόλο τη δέσμευση του οποιοδήποτε άλλου συναδέλφου όσον αφορά την ε, καταδίκη της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο για όλους. Και το θέμα που διακυβεύτηκε στην πρώτη ψηφοφορία δεν ήταν αυτό. Το θέμα μας ήταν θα τροποποιήσουμε ή όχι τα θέματα τα οποία είχαν ευρύτατα συζητηθεί. Γίνανε διάφορες συζητήσεις για το εάν κάποια θέματα ε, αμφιλεγόμενα θα περνούσαν. Ε, το πεδίο εφαρμογής, η περίοδος κράτησης, τα στοιχεία που αφορούν τις πτήσεις που αφορώνται ενδοκινοτικές προς τρίτες χώρες, υπερατλαντικές, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς χώρες και εδώ λαμβάνουμε υπόψη την ε, σοβαρή εγκληματικότητα, δεδομένου ότι δεν μιλούμε μόνο και για την τρομοκρατία. Ο στόχος της πρότασης δεν αφορά μόνο τρομοκρατικά χτυπήματα, αλλά και σοβαρή, σοβαρή εγκληματικότητα. Εγκλήματα τα οποία προβλέπονται και από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύνυψης. Δεδομένου ότι υπάρχουν κι άλλες μορφές εγκληματικότητας που στοχεύουμε εδώ. Κανείς λοιπόν εδώ δεν έχει το δικαίωμα να δυσπιστεί όσον αφορά τη δέσμευση κάποιου άλλου συναδέλφου όσον αφορά την ε, αγώνα που κάνουμε όλοι κατά της τρομοκρατίας. Ας κάνουμε όμως μια διευκρίνηση για την διαδικασία. Η απόρριψη της ε, ψηφοφορίας αφορά την εντολή διαπραγμάτευσης. Και αυτό ήταν το μόνο που μπορούσαμε να ψηφίσουμε, διότι θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο φάκελος αυτός, αυτό το θέμα το τόσο λεπτό, το PNR και το τόσο αντιφατικό, όπως φάνηκε και με σαφήν από τη συζήτηση, είναι ένα πεν, ένας από τους πέντε φακέλους που μπλοκαρίστηκαν μετά από τη διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι τις, ε, αυτό που λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από την απόφαση του Συμβουλίου να αλλάξει η νομική βάση του κώδικα που αφορά τα θέματα κανονισμών Schengen. Έτσι λοιπόν Λήφθηκε αυτή η απόφαση από το Συμβούλιο, αντιδράσαμε και η διάσκεψη των Προεδρών αποφάσισε να μπλοκάρει πέντε φακέλους. Τον ε, κώδικα για τα σύνορα, την αξιολόγηση, το εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, όλα αυτά στα πλαίσια του Σέγγεν, το PNR και πέντε μπλοκ πέντε φάκελοι μπλοκαρίστηκαν. Αυτό λοιπόν το πακέτο έχει μπλοκαριστεί από την διάσκεψη του Πρόεδρου, που είναι το μόνο ενδεδειγμένο και υπεύθυνο σώμα να αλλάξει αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένω να παραπέψουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια, αλλά και εδώ η απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο από τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Αν υπάρχει πλειοψηφία μεταξύ ημών, θα αποστείλω επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων ώστε να θέσω το όλο θέμα σε αυτούς την διάσκεψη των Προέδρων οι οποίοι θα λάβουν την απόφαση ουσίας. Αλλά η διάσκεψη των Προέδρων, επαναλαμβάνω, είναι το όργανο το οποίο θα ξεμπλοκάρει το φάκελο αυτό. Μέχρι τότε δεν μπορεί να γίνει καμία ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί αυτών όλων των μπλοκαρισμένων φακέλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη αποφασιστεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω. Δηλαδή αυτή είναι η υπόδειξή μας όσον αφορά τη διαδικασία, εάν συμφωνείτε. Ο κύριος Βέμπερ. Να πω όλα πολλά, κύριε Πρόεδρε πως το ΕΛΚ εξακολουθεί να θεωρεί πως έπρεπε να έχει γίνει η τελική ψηφοφορία. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια το θέμα του backloading για το διοξείδιο του άνθρακα. Έγινε συζήτηση επί της ουσίας και ε, ψηφοφορία επί της ουσίας και μετά η τελική ψηφοφορία. Δύο διαφορετικές ψηφοφορίες. Έτσι γίνεται και στην Ολομέλεια. Και έτσι νομίζω πρέπει να γίνει και στην Επιτροπή. Αλλά αυτό είναι ένα ε, διαδικαστικό ζήτημα που είναι ανοιχτό. Θα ήθελα, ε, όπως είπατε και εσείς πράγματι, να πάει το ζήτημα στην διάσκεψη των Προέδρων και να σας παρακαλέσω επιπλέον. Γνωρίζουμε όλοι πως είναι σημαντικό το θέμα και ευαίσθητο. Και πρέπει όταν μια μεγάλα ομάδα θέτει ζητήματα διαδικασίας και δεν βγάζω επιχειρήματα από το κεφάλι μου σας ανέφερα άρθρα του κανονισμού. Όταν υπάρχουν λοιπόν ανοιχτά τέτοια ζητήματα, το εάν επιτρέπεται δηλαδή μια επιτροπή ή όχι να κάνει κάτι, νομίζω να τα αξιολογήσει η αρμόδια επιτροπή, η ΑΦΚΟ. Όταν υπάρχουν ζητήματα ερμηνείας του κανονισμού, η αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει, νομίζω, το ζήτημα αυτό να ξεχαρίσει οριστικά για να ισχύσει και για άλλε περιπτώσεις, το αν είναι δυνατόν δηλαδή να απορρίπτουμε νομοθετικές εκθέσεις. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρο να υποβληθεί το θέμα αυτό στην διάσκεψη των Προέδρων για να αντιμετωπιστεί σωστά. Με πρόλαβε ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Εδώ πέρα δεν επρόκειτο για κάποια α, οριστική ψηφοφορία. Ήταν μια τροπολογία αυτή η οποία ψηφίστηκε. και πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Έτσι είναι η διαδικασία και αυτό το οποίο ζητάω είναι να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σήμερα επί του κειμένου αυτού. Μπορείτε να δείτε και τον κανονισμό, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε απλά ψηφίσει μία τροπολογία η οποία βεβαίως σημαίνει πως οι υπόλοιπες καταπίπτουν, αλλά το κείμενο συνολικά δεν έχει ψηφιστεί. Και να σας πω πως δεν ήταν αυτή η τελική ε, ψηφοφορία. Συγγνώμη, ο κύριος ε, Βοητσόφσκι έχει ζητήσει το λόγο πρώτος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πραγματικά μου κάνει εντύπωση το ότι ε, υπάρχουν τόσα διαδικαστικά προβλήματα, ενώ, ενώ λογικά υπάρχει ένας ξεκάθαρος κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προβλέπει ψηφοφορία στην Ολομέλεια, το άρθρο 56. Το άρθρο 56 προβλέπει ένα τέτοιο ενδεχόμενο όταν έχει απορριφθεί μια πρόταση από μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η Επιτροπή μας απέρριψε την έκθεση αυτή, αλλά θα πρέπει να ψηφιστεί η έκθεση αυτή στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Και αφού γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής στην Ολομέλεια, η Επιτροπή μας ή θα διατηρήσει το ψήφισμα ή θα το απορρίψει. Πάντως, η διαδικασία περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια στον κανονισμό μας. Η δική μας ψηφοφορία δεν αποτελεί το τέλος της ιστορίας. Η πρόταση αυτή, επαναλαμβάνω, πρέπει να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο προκύπτουν τόσα πολλά διαδικαστικά προβλήματα. Εν προκειμένου, οι κανόνε είναι ξεκάθαροι. Κυρία Ρομέρο, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η ψηφοφορία που έγινε καταρχήν δεν θα έπρεπε να μας οδηγήσει στο να μπούμε στην ουσία του όλου θέματος της πρότασης. Τι θέλω να πω, ότι η δική μου ομάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα εάν πάει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Είναι θέμα διαδικασίας και τήρησης των κανονισμών. Το ΕΛΚ όμως, προφανώς, δεν έχει συνηθίσει να χάνει ψηφοφορίες. Εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχασε την ψηφοφορία, προφανώς υπάρχουν διαδικασίες νόμιμες οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν ξέρουμε αν διάσκεψη των προέδρων ή κάποια άλλη διαδικασία θα βγάλει το διατάφτα. Αλλά υπάρχουν μέσα ε, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε όταν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, όποιος και αν είναι υπεύθυνο για την λήψη αυτή τη απόφαση, α το αποφασίσει. Αλλά μην συνεχίσουμε τη συζήτηση επί τη ουσία μία πρόταση η οποία απορρίφθηκε με το καλημέρα σα, με την πρώτη ψηφοφορία. Το δεχθεί το ΕΛΚ και από εκεί και μετά α γίνει η συζήτηση επί τη διαδικασία. Αλλά θα πρέπει κάποιο υπεύθυνο, αρμόδιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει πώ εφαρμόζει σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση ο κανονισμό. Ευχαριστώ. Κύριο Όλμπρεχτ. Νομίζω πως πρέπει νομίζω να δεχτούμε πως ελήφθη μια απόφαση. Όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, επαρκεί νομίζω αυτή η απόφαση ε, για την απόρριψη. Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη ε, ψηφοφορία γιατί θα έχουμε επανάληψη του ίδιου πράγματος. Το εάν θα πάει τώρα στην Ολομέλεια ή όχι. Θα έλεγα ας το κρίνουν ε, οι υπηρεσίες να το εξετάσουν αλλά νομίζω σήμερα έχουμε τελειώσει. Ελήφθη η απόφαση για απόρριψη. Οι συντονιστές των μεγάλων πολιτικών ομάδων από το ΕΛΚ και το Σοσιαλιστές θέλουν να πάρουν το λόγο για να αποσαφηνίσουν την κατάσταση και θα ολοκληρώσουμε όμως μετά τη συζήτηση. Κυρία Μάτιο πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ψηφίσαμε την τροπολογία απόρριψη, αλλά δεν ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά τώρα την νομική κατάσταση και κανείς μας, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι δήμονα σε θέματα διαδικαστικά και η κυρία Ρομέρο Λόπες θεωρώ ότι έχει δίκιο κάθε φορά που αφισβητείται μια απόφαση, η νομική κατάσταση δεν είναι σαφής, προβλέπεται μια διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ζητήσουμε από τα αρμόδια όργανα μια αποσαφήνιση. Δεν νομίζω ότι πρόκειται εμεί σήμερα να καταλήξουμε σε μια λογική απόφαση, επομένω για ποιο λόγο να μην παραπέμψουμε το όλο ζήτημα στους, στις των συντονιστών και να δούμε εκεί αν θα απευθυνθούμε στη νομική υπηρεσία ή στη γραμματεία για να διερευνήσουν περισσότερο τους υφιστάμενους κανονισμούς. Έχουμε και άλλες συναντήσεις και σήμερα και αύριο και έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει λόγος να αποφασίσουμε τώρα. Η κυρία Ματιού. Κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε την τροπολογία πόλη, αλλά δεν νομίζω ότι τελειώσαμε την ψηφοφορία και πιστεύω ότι θα πρέπει να την ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Ήταν σαφέστατα τα αποτελέσματα της ψηφοφορία. Ναι, αλλά αφορούσαν μια τροπολογία, λέει η κυρία Ματιό, και δεν νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Πρέπει να προχωρήσει ο πρόεδρος για να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία. Mr. Moraes, the coordinator for the about the procedure, the way... Για την ε, διαδικασία, πώς θα προχωρήσουμε κύριε Μωράης. Από βλέπω ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας σήμερα. Τελειώσαμε. Εκφράσαμε την άποψή μας. Ακούσαμε τι είπε και ο εισηγητής και άλλοι συνάδελφοι. Και από ό,τι ελέγχθη, ίσω σύμφωνα με το άρθρο 56 πάει στην Ολομέλη αλλά ούτω ή άλλω θα πρέπει η νομική υπηρεσία να διευκρινίσει το όλο θέμα. Από όσο κατανοώ, θα πρεπει η νομικη υπηρεσια να διευκρινισει το ολο θεμα απο οσο κατανοω μπορεί ενδεχομένω να πάει στην Ολομέλεια. Και αν ε, αποφασίσει ότι πρέπει να επανέλθει στην Επιτροπή μας, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιοι συμβιβασμοί μεταξύ των επικεφαλίστων ομάδων για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι έτσι εγώ καταλαβαίνω τα πράγματα. Έτσι εμείς το κατανοούμε όσον αφορά τη διαδικασία. Δεν εξαρτάται οτιδήποτε γίνει από πολιτική απόφαση θα λάβουμε σήμερα, εξαρτάται από τι προβλέπει η διαδικασία και ο κανονισμός. Αυτό που θα θέλαμε να συμβεί ως ομάδα είναι να διευκρινιστεί το συντομότερο δυνατό του τι ακριβώς διαδικασία θα ακολουθήσουμε εφ' εξής και να αρχίσουμε την εφαρμογή της. Αυτά. Σας ευχαριστώ όλους. Είχαμε μια διεξοδική συζήτηση. Ας προσπαθήσω να συνοψίσω εγώ τώρα. Καταρχάς, νομικές διευκρινήσεις. Σύμφωνα με μια νομική αρχή που ισχύει για όλες τις καταστάσεις, προβλέπεται το ακόλουθο. Δεν μπορεί ένα νομικό σώμα να ταχθεί κατά των νομικών του αποφάσεων. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσαμε, επομένως, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να ψηφίσουμε περαιτέρω, γιατί δεν μπορούμε να έρθουμε εμεί σε αντίφαση με την αρχική μας την απόφαση, με την αρχική μας την νομική βούληση, την οποία εξέφρασε η Επιτροπή αυτή. Άρα δεν προβλέπεται περαιτέρω ψηφοφορία. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση να μην περιμένατε την, το αποτέλεσμα αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή έχει ληφθεί μια νομική πολιτική απόφαση, δεν προβλέπεται συνέχιση της ψηφοφορίας πρόκειται για μία ψηφοφορία προς ανατολισμού όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, έχουμε το επόμενο στάδιο, δηλαδή την Ολομέλεια. Πάμε δηλαδή στην Ολομέλεια, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει αντίδραση, αντίθεση με την πρόταση του κυρίου Βέμπερ. Η διάσκεψη των Προέδρων έχει λάβει ήδη μία απόφαση ότι καμία ψηφοφορία στην Ολομέλη δεν μπορεί να γίνει για κανέναν από τους πέντε φακέλους που έχουν μπλοκαριστεί. Απόφαση η οποία ελήφθη για τη δέσμη Σέγγεν μετά την αλλαγή της νομικής βάσης του κώδικα συνόρων Σέγγεν. Απόφαση που πήρε το Συμβούλιο πριν από κάποιους μήνες. Εμείς θα γράψουμε λοιπόν προς την διάσκεψη των Προέδρων, θα υποβάλουμε το αίτημά μας και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς από νομικής πλευράς μπορούμε να παραπέμψουμε την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια. Που άλλωστε είναι το τελευταίο αυτό σώμα το οποίο μπορεί να αποφανθεί για τα ζητήματα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα προηγούμενο σε σχέση με τον τρόπο που διεξήχθη σήμερα η συζήτηση και αναφέρομαι στο νομοθετικό πακέτο όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα για την εγκληματικότητα, όπου ο κύριος Κίρχοπ ήταν και πάλι συγητής, απερίφθη σε μία πρώτη φάση, άρα δεν έγινε καμία άλλη ψηφοφορία για τις επιμέρους τροπολογίες του φακέλου αυτού, Έγινε μάλιστα μία δήλωση από την Επιτροπή με απόρριψη και αποφασίσαμε τότε ότι δεν θα γινόταν καμία άλλη ψηφοφορία. Τελεία και παύλα είχαμε πει τότε για το συγκεκριμένο κοινοφάκελο. Έτσι είχαμε λειτουργήσει τότε με την έκθεση αυτήν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ολομέλεια πάλι θα είχε τον τελευταίο λόγο. Επομένως, ας ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και για αυτή την έκθεση. Ας παραπεμφθεί η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια και εκεί πέρα θα δοθεί μια λύση. Μπορεί προσωρινά να ολοκληρώνεται εδώ η διαδικασία. Έχουμε άλλωστε και την συνεδρίαση των συντονιστών αυτή τη στιγμή. Κύριε Φώσα, τελευταία όμως παρέμβαση παρακαλώ. Να Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, να ακούσουμε τον κύριο Φως. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Το ζήτημα του μπλοκαρίσματος δεν έχει σχέση με το τωρινό. Το ερώτημα είναι εάν με αυτή τη μία ψηφοφορία χωρίς τελική ψηφοφορία μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί νομικά. Να σας πω, Οπωσδήποτε έχει σχέση γιατί ακριβώς η απόφαση που ελήφθη ομόφωνα από τη διάσκεψη των Προέδρων ήταν πως δεν θα υπάρξει ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ακριβώς αυτή ήταν η απόφαση μου. Το είπαν ξεκάθαρα πως ε, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε επί των θεμάτων, αλλά δεν θα λάβει χώρα ψηφοφορία στην Ολομέλεια εκτός εάν και μέχρι να ε, ληφθεί συνολική απόφαση για τον μπλοκάρισμα του θέματος όλου του πακέτου των πέντε αυτών θεμάτων ε, από τη διάσκεψη των Πρόεδρων. Μου το είπαν ξεκάθαρα. Οπότε ας το υποβάλουμε στη διάσκεψη των Πρόεδρων και να δούμε τι θα γίνει με την